Ήταν μια γενναία γυναίκα, μια σπουδαία δημοσιογράφος. Και άσκησε αυτό το λειτουργήμα για να ερευνήσει, να ανακαλύψει την αλήθεια τα πραγματικά περιστατικά χωρίς κανένα φόβο για κανέναν. Κανέναν φόβο για να φτάσει μέχρι το τέλος. Για να κάνει το καθήκον της. 30 χρόνια σταδιοδρομίας. Ποτέ δεν έχασε την ορμή της. Προσπάθησε να ρίξει φως στα σκοτάδια και προσπάθησε να είναι πιστή στους αναγνώστες της. Μόνος σε αυτούς θεωρούσε ότι οφείλει να λογοδοτεί. Πάνω από 20.000 άρθρα έγραψε και ρέγαψε τις καταχρήσεις της εξουσίας, διαφθορά και κακοδιοίκηση. Όπως κάθε πραγματικός δημοσιογράφος. Αυτή ήταν πρωτοπόρα, ήταν στρατιώτες στην πρώτη γραμμή για την υπεράσπιση των αξιών μας. Και μόνο ένας ελεύθερος και ανεξάρτητος τύπος μπορεί να μας δώσει την ευκαιρία να προστατεύσουμε την δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την ελευθερία έκφρασης. Όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα που είναι το θεμέλιο της ευρωπαϊκής οικοδόμησης, θεμέλια του ίδιου του πολιτισμού μας. Είναι πολύ παραπάνω Ευρωπαϊκή Ένωση από μια τραπεζική ένωση, από μια νέα αγορά. Είναι ο καθρέφτης των αξιών μας, της ε, προσωπικής ατομικής αξιοπρέπειας και ελευθερίας για να μπορέσουμε να την προστατεύσουμε κάθε μέρα. Θα πρέπει να επιβεβαιώνουμε την ανεξαρτησία του τύπου. Είμαι περήφανος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντοτε και δυναμικά στρατεύεται προς αυτό το μέτωπο. Η δολοφονία της Δάφνης δεν θα πρέπει να μείνει ατιμόρυτη. Άρα θα πρέπει έτσι να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τους δημοσιογράφους, θα πρέπει να υπάρχει προστασία ε, από τη δικαιοσύνη πρώτα-πρώτα εδώ στην Ευρώπη και προσδοκώ από τις ε, αρχές της Μάλτας να καταβάλουν πάσα την αντιπροσπάθεια ούτως ώστε να πέσει άπλα το φως πάνω σε αυτό το έγκλημα και θα πρέπει να ερευνήσουν κάθε πιθανότητα. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο και η Europol να εμπλακεί στα πλαίσια μιας διεθνούς ερεύνης. Οπότε θα πρέπει και πάσα διοκτική αρχή να μπορέσει να βοηθήσει ούτω ώστε να συλληφθούν και να καταδικαστούν οι ένοχοι. Και αυτού του είδους η διεθνής συστράτευση αναφέρθηκε στην τελευταία συνάντηση αρχικών κρατών και κυβερνήσεων στην Ένωση. Έδωσε το παράδειγμα προς μίμηση η Δάφνη και αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Γι' αυτό, χθες το απόγευμα, το γραφείο της Προεδρίας απεφάσισε να ονομάσει Δάφνη Καρουάνα Γκαλίτσε την αίθουσα τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Έχουμε την οικογένειά της εδώ που παρακολουθεί την Ολομέλεια, τον σύζυγο, τα τρία τέκνα. Οπότε και θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για τις χιλιάδες μελτές οι οποίοι κατέβηκαν στο πεζοδρόμιο την Κυριακή για να πούν το πόσο έχουν αισθανθεί για αυτή την υπόθεση και αυτοί προσωπούν χιλιάδες Ευρωπαίων. Αυτό το χειροκρότημα αγαπητή οικογένεια της Δάφνης αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πάψει να ασχολείται με την δολοφονία της γυναίκας, της μητέρας της δικής σας μέχρι ότου αποκαλυφθεί η αλήθεια. Δεν θα σταματήσουμε να ασχολούμαστε μέχρι ότου ανακαλυφθούν οι ένοχοι αυτής της δολοφονίας. Και τώρα παρακαλώ για ενός λεπτού σιγή προς τιμήν αυτής της γυναίκας. Στη μνή της Δάφνης Καρόνα Γαλίτσια. Ο κύριος Κόρβιν Μίκε για διαδικαστικό. Η Μαλτέζικη κυβέρνηση ε, ζήτησε να υπάρξει, έχει θέσει ένα εκατομμύριο αμοιβή για αυτούς που θα βοηθήσουν να βρεθεί ο ένοχος του κλίματος αυτού. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφε να περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες για την έκθεση ΡΙΚΕ. Η κυρία Σνάλφος για διαδικαστικό παρακαλώ. Μόλις αποτίσαμε φόρο τιμής στην κυρία ε, Καρουάνα Γαλίσια. Ήταν αναγκαίος αυτός ο φόρος τιμής, αλλά ο φόρος τιμής ο πραγματικός θα ήταν ε, να κάνουμε τα ε, ε λόγια δράση εδώ και ε, ε, σε λίγο καιρό θα ψηφίσουμε μία έκθεση για αυτούς οι οποίοι καταγγέλνουν τα κακό κείμενα. Παρακαλώ να καταψηφίσετε τις τροπολογίες που προσπαθούν να τους εμποδίσουν.